που έγιναν σε πνεύμα συνεργασία που ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. The Έληξε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι η έκθεση του κυρίου Κατσμάρεκ με θέμα τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής. Έχετε τέσσερα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση που παρουσιάζω σήμερα έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης εξωτερικής βοήθειας. Είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται χρόνια και ουσιαστικά περνάει το επίκεντρο της διαχείρισης από την έδρα στις Βρυξέλλες στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωση στις δικαιούχες χώρες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος λοιπόν περιλαμβάνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη εφαρμογή, ταχύτερη εφαρμογή και καλύτερη διαχείριση. Γι' αυτό και συμμετείχε στη διερεύνηση η Επιτροπή Κοκομπό. Ακόμη πρέπει να είναι καλύτερη ποιότητα της βοηθείας που παρέχεται στην χώρα για την οποία πρόκειται. Σίγουρα συμφωνείτε ότι μια αποκεντρωμένη προσέγγιση έχει διάφορα πλέον εκτήματα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο κοντά στους δικαιούχους. Λειτουργικά αυτό είναι πιο αποτελεσματικό και έχουμε καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων των διαφόρων δωρητών. Ταυτόχρονα έχουμε και λογοδοσία ε, σε σχέση με τα τοπικά ε, τους τοπικούς οργανισμούς. Βεβαίω η αποκέντρωση δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Χρειάζονται και πρόσθετες δράσεις για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Η βοήθεια που διοικείται αποκεντρωμένα καλύπτει ευρύ φάσμα. Ουσιαστικά το φάσμα είναι υπερβολικά ευρύ, γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε το συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούχων ε, κρατών και φορέων εφαρμογής. Θέλουμε καλύτερη κατανομή των ε, δράσεων ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να προχωρά και να βελτιώνει την αποτελεσματική η αποκέντρωση επίσης μειώνει το κόστος της ε, βοήθειας που παρέχεται. Είναι καλό αυτό, αλλά δεν είναι η μέθοδος για τη μείωση ε, των στοιχείων κόστους. Ακόμη χρειαζόμαστε υποστήριξη του προϋπολογισμού ώστε να επικεντρώνεται περισσότερο στις ανάγκες της χώρας στην οποία παρέχουμε τη βοήθεια. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα. Έχουν αλλάξει οι ομάδες, ε, αλλάζουν πολύ γρήγορα οι ομάδες που εργάζονται, οι ομάδες τελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται για τα θέματα αυτά επιτόπου. Γι' αυτό ζητούμε από την Κομισιόν να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία ώστε όλες αυτές οι δραστηριότητες να έχουν τη σωστή διαχείριση. Μας ανησυχεί ακριβώς αυτή η γρήγορη ανανέωση του προσωπικού που ουσιαστικά δεν αφήνει την εμπειρία να δημιουργηθεί. Ακόμη, έχουμε, θέλουμε να έχουμε συνοχή μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να επαληθεύονται τα αποτελέσματα. Είμαι πεπισμένος ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Ανάπτυξης πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στο θέμα της μείωσης της φτώχειας, ώστε να εκκριζωθεί τέλος πάντων η φτώχεια. Είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ακόμη, ούτε η Κομισιόν, ούτε τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την κρίση σαν αιτιολόγηση, σαν επιχειρηματολογία για να ε, επιδιώκουν περισσότερα με λιγότερα, διότι έτσι θα έχουμε χαμηλότερη στελέχωση των αντιπροσωπιών. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Και τώρα περνάμε στο Catch the Eye. Δύο μιλητές, ο κύριος Μπασέκου πρώτος. Κυρία Μπαζέκο, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική και στηρίζει τις θεσμικές αλλαγές οι οποίες οφείλονται στην συνθήκη της Λισαβόνας και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που αποκεντρώνει ένα μέρος της πολιτικής μας. Η διαχείριση της εξωτερικής βοηθείας από την αποστολή θα είναι μια καλύτερη λύση λόγω άμεσης επαφής με τον ε, τοπικό πληθυσμό και θα, υπάρχει, ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση για τη διαχείριση αυτών των πόρων. Θα χρειαστεί να υπάρξουν νέες νέα καθήκοντα, θα υπάρξει αποκέντρωση. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε τις νέες προτεραιότητες και που υπάρχουν επικαλύψεις. Στηρίζω τον λόγο, ε, ρόλο που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέρη. Η κυρία Φερέιρα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποτελεσματικότητα της βοήθειας στην ενίσχυση είναι ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας. Αυτό το θέμα ξεπερνάει τις πτυχές ε, ε, διαχείρισης από την Επιτροπή. Όπως είπε ο εισηγητής, χρειάζεται μία συνοχή μεταξύ των τομεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων της ενίσχυσης είναι απαραίτητο οι ενισχύσεις να λάβουν υπόψη τις αρχές της χώρας, τις κοινωνικές οργανώσεις και αυτό σε, ό,τι αφορά την εφαρμογή των πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να καθορίζει αλλά να στηρίζει. Θα πρέπει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες των υπονάπτυξη χωρών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεργασία ε, μεταξύ των νότιων χωρών. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες των υποανάπτυξη χωρών και όχι να διαιωνίζεται η εξάρτησή τους. Ένα σημαντικό μέρος των ενισχύσεων επιστρέφει στις χώρες προέλευσης για την γιατί αγοράζουν οι υπηρεσίες από τις ε, ε, χώρες δωρητές. Ευχαριστώ πολύ ο Επίτροπο Βαντόφσκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίω συμφωνούμε με την έκθεση του κυρίου Κασμάρη καθώς και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που μα δείχνει πώς ακριβώς ότι η αποκέντρωση επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Και πιστεύω ε, ότι ε, ε, η βοήθεια φτάνει πιο εύκολα στους δικαιώκους. για να μπορέσουμε να εξετάσουμε να καταλάβουμε το δυναμικό αυτής ε, της αποκέντρωσης θα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το θέμα το προσωπικό και εκεί χρειάζεται συνεργασία μεταξύ του, μέσα στο κοινοβούλιο. Βεβαίως θα, θα πρέπει πρέπει να αναλάβουμε την υποχρέωση να βελτιώσουμε τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του κυρίου Χασμάρα και του, ε, της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των ενισχύσεων της βοήθειας. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε στρώσουμε την προσοχή μας εκεί που πραγματικά χρειάζονται και εκεί που εντοπίζονται επιπρόσθετες ανάγκες, όπως για παράδειγμα στην Αφρική. Όπως αναφέρθηκε στο θέμα της εναλλαγής, αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα από τη στιγμή που το 40% των υπαλλήλων είναι συμβασιούχοι με συμβόλαια τριετή και η αύξηση αυτού του ποσοστού θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στο μέλλον. Συνεπώς για να αμβλύνουμε το πρόβλημα των συμβατησιούχων και την εναλλαγή των εργαζομένων ε, ε, ε, δίνουμε συμβάσεις στις αντιπροσωπίες μόλις περάσει η περίοδος της σύμβασης και θα επιθυμούσαμε να δίνονται συμβάσεις εξαετής και ο συνάδελφος και βεβαίω ζητάμε το Κοινοβούλιο υποστηρίξει τι προσπάθειέ μα σε αυτό το μέτωπο. Σε, η σχέση με τις εξωτερικές υπηρεσίες, βεβαίω πρόκειται για νέε υπηρεσίε. Ε, θα πρέπει να γίνει ένας καταμερισμός της εργασίας και υπάρχει βεβαίως η ευθύνη των επικεφαλής των αντιπροσωπιών οι οποίοι δεν είναι μόνο οι υπεύθυνοι ε, ε, γενικά αλλά και υπεύθυνοι για τη ροή των πραγμάτων αλλά είμαστε εμείς ο, ο επίτροπο ο Επίτροπος είναι απόλυτα υπόλογος στο Κοινοβούλιο και βεβαίως η από κέντρωση είναι μια θετική εξέλιξη. και Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και τις ε, συμβουλές που ε, ε, παρατίθενται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πέρα στη συζήτηση, σε ψηφοφορία αύριο στις 12. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι διακόπτουμε για δύο λεπτά και μετά συνεχίζουμε.